Dear uh, welcome. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε στην συνεδρίαση συγκρότησης ε, Σώμα της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ρόλος του απερχόμενου Προέδρου είναι να προεδρεύσει αυτή τη συνεδρίαση. Κυρίσω λοιπόν την έναρξη της συνεδρίασης. Όπως ε, θα γνωρίζετε, σκοπός της συνεδρίας αυτής είναι να εκλέξουμε τον ή την Πρόεδρο και μέχρι τέσσερις αντιπροέδρους δυνάμει του άρθρου 204 του ιστορικού κανονισμού η σειρά της ψηφοφορίας έχει ως εξή πρώτα εκλέγουμε τον πρόεδρο και μετά τους αντιπροέδρους να σας ανακοινώσω επίσης τα ονόματα των αναπληρωτών που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία και να ρωτήσω αν πρόκειται να υπάρξουν αλλα... ότι σε... να πω ότι σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές αργότερα θα ήθελα οι πολιτικές ομάδες να με ενημερώσουν πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Έχουμε τον κύριο Κούτσεφ που αντικαθιστά τον κύριο Ράντιεφ και την κυρία Σπινέλη που αντικαθιστά τον κύριο Χρυσόγωνο. Σωστά. Ας προχωρήσουμε τώρα στην εκλογή του Προέδρου ή της Προέδρου. Έχουμε φτάσει, έχει επιτευχθεί απαρτία, διότι τουλάχιστον ένα τέταρτο των μελών ε, αποτελούν την απαρτία, δηλαδή τουλάχιστον 7 μέλη της Επιτροπής Γιούρη. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω τις προτάσεις για τον Πρόεδρο. Κύριε Ρέγνερ, ε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θέλω να πω ότι λυπάμαι. Ένα από τα μέλη μας, ο κύριος Γκασπάρε, έχασε το τρένο και προσπαθεί να έρθει όσο, ε, προσπαθούμε να βρούμε όσο το δυνατόν συντομότερο τον αναπληρωτή του. Οπότε, ε, πέντε λεπτά αν μπορείτε να περιμένετε. Εννοείται να τον περιμένουμε. Θα ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Ξέρετε, η, η σύνθεση της Επιτροπής είναι τέτοια μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο κύριος Φώσης, ζητάει το λόγο. Λοιπόν, για τις προτάσεις. Το ΕΛΚ προτείνει τον Παύλ Σβόμποντα Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Δέχομαι την πρόταση. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι παρακαλώ. Άλλες υποψηφιότητες προτείνονται. Όχι. Θέλει κανείς να γίνει μυστική ψηφοφορία. Όχι. Ωραία, μπορούμε διαβοής. Ε, I Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για την εμπιστοσύνη σας και ελπίζω να συνεχίσουμε στην Επιτροπή μας όχι μόνο εργαζόμεθα αποτελεσματικά αλλά και φιλικά. Ευχαριστώ λοιπόν. Οπότε τώρα να εκλέξουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο. δεν έχει αλλάξει ο κατάλογος των ε, αντιπροματικών που παρευρίσκονται και απαρτία πάντα έχουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, υποψηφιότητες για τον πρώτο αντιπρόεδρο, η κυρία Ρέγνα. Η κυρία Λίντια Γκέριγκα Ευχαριστώ πολύ. Άλλες προτάσεις. Δεν βλέπω. Κυρία Γκέρνια, δέχεστε. Ευχαριστώ πολύ. Είστε τακτικό μέλος Επιτροπής μας. Υποθέτω ότι έχετε υποβάλει την δήλωση ε, περιουσιακών στοιχείων. Θέλει κανείς να υπάρξει μυστική ψηφοφορία. Όχι.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 Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Ζωμαρί Καβαντά στο όνομα της ομάδας Άλντ. Μάλιστα ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόταση. Υπάρχουν άλλες προτάσεις. Όχι. Ο κύριος Καβαντά συμφωνεί. Συμφωνείτε πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι έχετε συμπληρώσει τη δήλωση σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα. Είναι μια προϋπόθεση αυτή. Πολύ ωραία. Θέλει κάποιο μυστική ψηφοφορία. Όχι. Ωραία. Ας ψηφίσουμε διαβοής λοιπόν. Συγχαρητήρια κύριε Καβαντά. Παρακαλώ έλατε κι εσείς εδώ στο Προεδρείο. We can, we can proceed with uh, the election of the third uh, vice chair. Και τώρα θα εκλέξουμε τον τρίτο αντιπρόεδρο. Υπάρχουν υποψηφιότητες. Ευχαριστώ Πρόεδρε να προτείνω ως υποψηφίο τη συναδελφό μας Λάουρα Φεράρα. Uh, thank you very much. Μάλιστα, ευχαριστώ. Η κυρία Φεράρα συμφωνεί. Άλλες υποψηφιότητες δεν υπάρχουν. Ζητεί κανείς μυστική ψηφοφορία. Όχι. Η κυρία Φεράρα φαντάζομαι έχει και αυτή συμπληρώσει τη δήλωση για τα οικονομικά συμφέροντα. Πολύ ωραία διαβοής λοιπόν. Εκλέγεται η κυρία Φεράρα. Congratulations, Συγχαρητήρια. Παρακαλώ πάρτε και εσείς θέση. And we have uh, the last... Και έχουμε πλέον την εκλογή ε, της τέταρτης και τελευταίου αντιπροέδρου, κυρία Ρέγνερ. Προτείνω την κυρία Μάντι Ντελβό η κυρία Ντελβό συμφωνεί, συνενεί, πολύ ωραία και εσείς θα έχετε συμπληρώσει τη δήλωση, τη γνωστή, πολύ ωραία, έτσι ελπίζετε μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, δεν ζητεί κανείς μυστική ψηφοφορία, όχι. Διαβοής λοιπόν. Congratulations. Συγχαρητήρια κυρία Ντελβό. Πάτε και στη θέση παρακαλώ εδώ μαζί μας. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το καθήκον μας. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα τα πούμε αύριο στην τακτική... Α, συγγνώμη, την ερχόμενη εβδομάδα. Την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, στην συνεδρία της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ.